Ευχαριστώ. Η συζήτηση θα συνεχιστεί, ε, η συζήτηση έληξε και ε, η ψηφοφορία θα είναι αύριο Πέμπτη. Η επόμενη έκθεση είναι ε, του κυρίου Μάνκα σχετικά με την τροποποίηση της κατάστασης προβλέψεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον προπολογισμό του 2010 και δίνω τον λόγο στον κύριο Μάνκα για τέσσερα λεπτά, τον εισηγητή. Κύριε εισηγητά, έχετε το λόγο. Κύριε Επίτροπε, αγαπητοί συνάδελφοι, όλοι γνωρίζουμε πολύ καλά ότι με κοινή προσπάθεια της Ένωσης θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις μεγάλες προκλήσεις του 21ου αιώνα όπως είναι οι κλιματικές αλλαγές και η μείωση των πόρων, παγκοσμιοποίηση και απειλές στην ασφαλεία μας. Για να αντιμετωπίσουμε τέτοιου είδους προβλήματα η Ευρώπη θα πρέπει να έχει στη διάθεσή της τα κατάλληλα μέσα και αυτά είναι διαθέσιμα και μέσω της συνθήκης της Λισαβόνας. Πέρυσι το Δεκέμβριο εγκρίναμε τον προϋπολογισμό των θεσμικών οργάνων για το 2010 και εξαιτία της εφαρμογής της συνθήκης της Λισαβόνας δεν έχει τελειώσει η διαδικασία έγκρισης του προϋπολογισμού και θα συνεχιστεί μέχρι τον Απρίλιο. Εξ αρχής η Ένωση θα πρέπει να έχει τους απαραίτητους πόρους για να εφαρμόσει τις νέες πολιτικές. Η συνθήκη της Λισαβόνας θα έχει και άμεση και έμεση επίπτωση στις υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στα άλλα εθεσμικά όργανα. Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η συνθήκη θα επιφέρει διεύρυνση του πεδίου της συναπόφασης και θα ισχύσει για το 95% του νομοθετικού μας έργου και πολλοί τομείς τώρα πλέον μπαίνουν εντός της διαδικασίας της συναπόφασης. Αυτό θα ενισχύσει και την εφαρμογή της διαδικασίας της ειδική πλειοψηφία και στο Συμβούλιο. Βεβαίως αυτό θα οδηγήσει και σε αύξηση γενικότερα της νομοθετικής δραστηριότητας και αυτό θα επηρεάσει και την δραστηριότητα του Ευρωκοινοβουλίου, πράγμα το οποίο θα απαιτήσει ενίσχυση της διοικητικής μας δυνατότητας. Η κύρια, ο, ο, ο σκοπός της αύξησης αυτής της πρικοδότησης έχει σκοπό να εξασφαλίσει ότι θα εκπληρώσουμε τα καθήκοντά μας με βάση τη συνθήκη του Λισαβόνα. Το 1998 το Ευρωκοινοβούλιο έχει θέσει το 20% του συνόλου των διοικητικών δαπανών τότε ως όριο. Το 2006 στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο μέχρι το 2013 το Ευρωκοινοβούλιο ενέκρινε αυτό το επίπεδο των δαπανών ως μέγιστο για τις διοικητικές δαπάνες. Από το 2006 οι δαπάνες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουν αυξηθεί και παρά όλα αυτά τα γεγονότα για το καθεστώς των μελών και τη συνθήκη όλα αυτά δεν τα έχουμε λάβει υπόψη στον υπολογιστό για το 20% ως όριο. Παρόλα αυτά η Επιτροπή προϋπολογισμού επέμεινε ώστε ο προϋπολογισμός του Ευρωκοινοβουλίου να μην υπερβαίνει αυτό το όριο και το επιτύχαμε αυτό. Συντάσσοντας τώρα τον ε, προϋπολογισμό του 2011 θα πρέπει προσεκτικά να καθορίσουμε τα μεγέθη για να έχουμε βιωσιμότητα μέσα στο μέλλον και ο καλύτερος τρόπος για να επιτύχουμε βιωσιμότητα του προπολογισμού θα πρέπει να δούμε τις βασικές ανάγκες Τώρα οι ομιλητές για, από τις πολιτικές ομάδες. Ο κύριος Φερνάντε. Ευχαριστώ αγαπητοί συνάδελφοι κυρία Πρόεδρε. Αυτό το διορθωτικό προπολογισμό απορρέει από τη θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας. Αναλαμβάνει νέα καθήκοντα το κοινοβούλιο, νέες ευθύνες και γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να έχει τα κατάλληλα μέσα για να ανταποκριθεί σε αυτή τη νέα Υπογραμμίζω ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες απαιτούν την καλύτερη δυνατή νομοθεσία από το Ευρωκοινοβούλιο. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει οι, τα μέλη, οι επιτροπές και οι πολιτικές ομάδες να διαθέτουν τα απαραίτητα μέσα. Τα νομικά μέτρα, τα μέτρα του προϋπολογισμού και η χρηστή διαχείριση περιλαμβάνονται σε αυτόν τον διορθωτικό προϋπολογισμό. Θεωρούμε επίσης ότι η εξοικονόμηση θα πρέπει πάντα να είναι παρούσα και αυτό ελπίζουν και οι πολίτες και την ώρα που συζητούμε αυτόν τον προορθωτικό προπολογισμό. Γι' αυτό λοιπόν επαναλαμβάνουμε την υποβολή ενός μηδενικής αύξησης προϋπολογισμού και θα δίνει περισσότερες πληροφορίες για τις πραγματικές ε, δαπάνες του Ευρωκοινοβουλίου. Χρειάζεται μακροχρόνιος προ... προγραμματισμός της πολιτικής ακινήτων για να έχουμε βιωσιμότητα του προπολογισμού και μειώσαμε το αποθηματικό για τα κτίρια κατά 4 εκατομμύρια ευρώ. Με τον τρόπο αυτό το γενικό επίπεδο του προϋπολογισμού είναι το 19,99% του αρχικού τμήματος του κεφαλαίου 5 που εγκρίθηκε με πρώτη ανάγνωση και εγκρίθηκε το ποσό αυτό. Είμαστε σίγουροι ότι τα μέσα αυτά θα μας επιτρέψουν να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των Ευρωπαίων πολιτών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τώρα ο κύριος Σοφέρ με ονόμα της Σοσιαλιστικής Ομάδας. Κύριε, κύριε συνάδελφοι, πρόκειται για πρακτικά μέτρα για να μπορέσει να λειτουργήσει σωστά το Κοινοβούλιο αφού τεθεί ενισχύει η συνθήκη της Λισαβόνας. Πρόκειται για μια συμφωνία 20 ετή ε, βάσει της οποίας ε, θα έχουμε 20% του κεφαλαίου 5. Ε, έχουμε υπερβεί τα όρια αυτά λόγω πολιτικής και το 2011 το περιθώριο αυτό θα το υπερβούμε αν δεν περιορίσουμε ορισμένες δαπάνες σημαντικά σε ορισμένα σημεία. Και ε, το λέω αυτό διότι οι ε, δαπάνες μας έχουν αυξηθεί περισσότερο από ό,τι άλλων περιοχών και επίσης θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι ορισμένα κράτη-μέλη μειώνουν το προσωπικό και τους μισθούς. Δεν μπορούμε εμείς να αυξάνουμε ε, το κοινοτικό προσωπικό συνεργαζόμαστε και με άλλα θεσμικά όργανα και το 1998 είχαμε συμφωνήσει εάν υπερβούμε το 20% να γίνεται σε ε, συζήτηση με το Συμβούλιο, πράγμα το οποίο όμως θα δημιουργήσει προβλήματα σε όλες τις δημοσιονομικές συζητήσεις και γι' αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη αυτό για το μέλλον. Τώρα ε, δίνω το λόγο στην κυρία Βέρτμαν για 1,5 λεπτό. Κυρίες και κύριοι, το, η συνθήκη της Λισαβόνας έχει ενισχύσει την Ευρωπαϊκή Ένωση προς όφελος των ε, Ευρωπαίων πολιτών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Με την αναβάθμιση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δημιουργούνται και μεγαλύτερες νομοθετικές υποχρεώσεις οι οποίες θα πρέπει να καλυφθούν από όλους τους ευρωβουλευτές κατά συνείδηση και θα ήθελα εδώ να αναφερθώ εις ε, τα θέματα της νομοθεσίας. Ε, διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μία συνεχώς μεγαλύτερη κρίση και πρέπει γι' αυτό να προσέχουμε πολύ τα δημοσιονομικά μας διότι είμαστε υποχρεωμένοι σαν κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι να διεκπαιρεώνουμε σωστά τα καθήκοντά μας και αυτά τα θέματα πρέπει να ληφθούν υπόψη. Ε, τώρα το λόγο έχει ο Γκαρίγκα Πολέντο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. απόδειξη της εμπιστοσύνης που τρέφουν τα μέλη του Κοινοβουλίου προς, την Επιτροπή Προϋπολογισμού είναι ότι έχουμε φτάσει να, ψηφίσουμε, να ψηφίζουμε εδώ τέτοια σημαντικά θέματα όπως είναι οι αποζημιώσεις των κοινοβουλευτικών βοηθών και είμαστε μόνο τέσσερις νοματέοι μες στην Ολομέλεια. Οι συντονιστές ε, του των Σοσιαλιστών και του ΕΛΚ βρισκόμαστε εδώ για να πούμε ότι συμφωνούμε με την αύξηση του προϋπολογισμού διότι δεν παραβιάζει τους ε, κανόνες που ε, ε, τους κανόνες λιτότητας που μόνοι μας θέσαμε το κοινοβούλιο είναι ένα ιδιόμορφο όργανο Ξέρουμε πάρα πολύ καλά και ο κύριος Φάρμ και εγώ ότι αν στην Σουηδία ή αν στην Ισπανία το κοινοβούλιο αύξανε τις ε, αρμοδιότητες που, που έχει τότε θα έπρεπε αντίστοιχα να αυξήσει και τον προϋπολογισμό του. Αυτό μας συμβαίνει και σε μας. Τώρα στο μέλλον εμείς θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει μία εφορία αυτών των δαπανών διότι θα πρέπει να συζητήσουμε και για την κτηριακή πολιτική και για την διοικητική πολιτική του Κοινοβουλίου. Το Προεδρείο του Κοινοβουλίου και η Επιτροπή Προϋπολογισμών είχαν κάποιες διστάμενες απόψεις αλλά τελικά ε, διότι το Προεδρείο προστατεύει τα συμφέροντα όλων των βουλευτών, η Επιτροπή Προϋπολογισμών ε, τους κανόνες, αλλά τελικά είχαμε έναν καλό συμβιβασμό. Ο κύριος Βόγκαν. Μιλώ εξ ονόματος των Σοσιαλιστών και Δημοκρατικών Όλοι αναγνωρίζουν την ανάγκη περαιτέρω πόρων μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας, όμως υπάρχουν ερωτήματα για την χρηματοδότηση αυτών των προτάσεων. Υπάρχουν και άλλα θέματα, παραδείγματος χάρη, εάν έχουμε περισσότερους πόρους για το προσωπικό, με τι βάση καταλήξαμε σε αυτή την απέτηση, έχουμε στοιχεία και αποδείξεις. Θα υπάρξει επιπλέον προσωπικό για τη γραμματεία και αυτό θα πρέπει να το μάθουμε. Αν δεχτούμε την επιπλέον βοήθεια χιλίων ευρώ το μήνα θα πρέπει να δούμε και το, τα άλλα κόστη για περαιτέρω χορογραφίων και θα έχουμε μια σφαιρικό κόστος για αυτό. Πρόεδρε, θα είναι δύσκολη η απόφαση για τα μέλη αύριο. Πάντα είναι αμφιλεγόμενο όταν ζητάτε από τον εαυτό σας νέους πόρους. Αν είχαμε τις πληροφορίες που είχαμε ζητήσει θα μπορούσαμε να λάβουμε πιο ενημερωμένοι τις αποφάσεις μας αύριο. Ο κύριος Γκερμπράντι. Ευχαριστώ πρόεδρε λόγω της προχωρημένης ώρας. μπορούμε να πούμε ότι ακόμη δεν είδε φως στον ορίζοντα ο προϋπολογισμός. Η Λισαβόνα μας έχει δώσει νέες αρμοδιότητες, άρα θα χρειαστούμε και περισσότερα κονδύλια και για τις ομάδες και για το κοινοβούλιο και για τα μέλη. Εγώ έχω αμφιβολίες όμως. Πιστεύω ότι μπορούμε και μέσα σε αυτόν τον προπολογισμό να εργαστούμε αποτελεσματικά ή όχι. Πολλά βήματα πρέπει να γίνουν. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα μέσα σε ένα χρόνο. Στο μέλλον θα συντηθούν αυξήσει με τις οποίες δεν θα συμφωνήσει η ομάδα μας. Ένα και μία και μοναδική αύξηση θα υπάρξει για μας που δεν μπορεί να επαναληφθεί του χρόνου. Ο κύριος Μαρινέσκου. Ευχαριστώ. Η νομοθετική αριστεία είναι σημαντική εδώ και πρέπει να βρούμε τρόπο να την επιτύχουμε διότι οι ε, δημοσιονομικές δυνατότητες που περιλαμβάνονται στις συνθήκες Λισαβόνας τώρα έχουν υιοθετηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μπορούν να ενισχύσουν το νομοθετικό ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και την ανάγκη προσθήκης περαιτέρων πόρων, διότι για να υπάρχει σταθερότης θα πρέπει να έχουμε μια καλή δημοσιονομική πολιτική και μια βραχυπρόθεσμη πολιτική όσον αφορά την κτηριακή πολιτική του Κοινοβουλίου. Νομίζω ότι θα έπρεπε να παραμείνουμε στο αρχικό πρόγραμμα, στο πολιετές πλαίσιο και στην δημοσιονομική πειθαρχία να διατηρήσουμε το παραδοσιακό επίπεδο του 20% και χαιρετίζω την συμφωνία να μην υπερβούμε αυτό το επίπεδο εδώ κατά τρόπον ώστε να υπάρξει αηφορία του προϋπολογισμού στα επόμενα έτη και γι' αυτό χρειάζεται μία ε, πολιτική η οποία θα είναι πιο αυστηρή. Θέλουμε διαφάνεια και περισσότερη πληροφόρηση όσον αφορά τα συνολικό, τις συνολικές δαπάνες της του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και τώρα έχω έναν ομιλητή μόνο για το Catch the Eye, τον κύριο Ρούμπι. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα στην ολοκλήρωση αυτής της συζητήσεως να σας πω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο αναλαμβάνει τις ευθύνες του και θα ήθελα εδώ να ευχαριστήσω το Προεδρείο διότι ευρέθη η δυνατότητα να κρατήσουμε αυτό το ανώτατο επίπεδο των 20% που είναι πολύ σημαντικό διότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε περίοδο οικονομικής κρίσεως με τα χρήματα των φορολογουμένων και συγχρόνως να κοιτάξουμε να καλύψουμε τις ανάγκες των Ευρωβουλευτών. Όσον αφορά τα 4 εκατομμύρια περικοπή από την κτηριακή πολιτική δεν πρέπει να ανησυχούμε διότι το Κοινοβούλιο είναι ένα από τα πιο σύγχρονα κτίρια σε αυτό τον κόσμο και ε, θα πρέπει εμείς να μπορούμε να δουλέψουμε σωστά προς όφελο των πολιτών. Ευχαριστώ και το λόγο δίνω τώρα στον κύριο Μάν και τον εισηγητή μας για δύο λεπτά. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα τώρα να ευχαριστήσω όλους εσάς για τις απόψεις σας και τη συνεισφορά σας για να βρεθεί μια λύση εντός της Επιτροπής. Σας υπενθυμίζω ότι στον προϋπολογισμό του 2010 έχουμε συμπεριλάβει συστημικά μέτρα για εξοικονόμηση πόρων και να μειώσουμε τις πιέσεις στους πόρους μας. περασμένο Οκτώβριο, κατά τη διάρκεια της συνδιαλλαγής, συμφωνήσαμε το Ευρωκοινοβούλιο να είναι αντικείμενο εσωτερικού ελέγχου και η ιδέα είναι να δούμε το εάν χρησιμοποιούμε τους σπόρους μας με τον βέλτιστο τρόπο. Θα χρησιμοποιήσουμε τη γνώση αυτή για να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητά μας. Μπορεί να υπάρχουν περισσότερα αποθυματικά στην καλύτερη χρήση της διερμηνίας ή στην τελεργασία. Αναμένουμε ότι και τα άλλα θεσμικά όργανα θα μας ενημερώσουν για το πώς θα χρησιμοποιήσουν όχι μόνο τις γλωσσικές δυνατότητες αλλά και τις δυνατότητες ενοικίασης, φωτοτύπησης κτλ. Είμαι πεπισμένος ότι οι εξοικονομήσεις θα επιτευχθούν με τον μεσοπρόθεσμη στρατηγική στην κτηριακή πολιτική που θα μας υποβάλει η διοίκηση του Κοινοβουλίου. Αναμένουμε σε μερικές μέρες να λάβουμε αυτή τη στρατηγική. Σας ευχαριστώ για την συνεργασία σας για άλλη μια φορά. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ λίγη η συζήτηση και αύριο 11.30 ώρα πέμπτη ε, θα γίνει ψηφοφορία. Αύριο θα είναι η επόμενη συνεδρίαση 25 ε, Φεβρουαρίου από τις 9.30 ως τη 1. Η έκθεση έχει 9 ε, μέχρι την